Καλώ ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι στην απογευματινή τελευταία μα συνεδρίαση πριν τι ε, πασχαλινές διακοπέ. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ το απόγευμα στην Επιτροπή μα, τον κύριο Φίλ Γουίν Owen. Καλώ ήρθατε κύριε Owen που είναι μέλος του πρότματος του ελεγκτικού συνεδρίου και θα μας παρουσιάσει την ειδική έκθεση. Πρόκειται για την ειδική έκθεση που αφορά τις δαπάνες, τις περιβαλλοντικές δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Θα μιλήσουμε για την ε, ανάγκη ε, αντιμετώπιση πρόκληση του μετριασμού των κλιματικών αλλαγών και των συναφών επενδυτικών ε, αναγκών σε τουλάχιστον 20% του ενωσιακού προϋπολογισμού για την περίοδο προγραμματισμού. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό, η έκθεση αναφέρει ότι μεταξύ άλλων οι τομείς της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, ανάπτυξης υπαίθρου δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη αλλαγή προς μία κλιματική δράση και εντοπίζει επίσης τον κίνδυνο να μην υλοποιηθεί ο στόχος του 20% των δαπανών για περιβαλλοντικές δράσεις. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν ο κ. Γουινόμεν τα πορίσματα της έκθεσης, της ειδικής αυτής έκθεσης του Ερεκτικού Συνεδρίου. Στη συνέχεια θα υποβάλουμε ερωτήσεις. Και μάλιστα ο τίτλος της έκθεσης είναι πολύ καλός. Η δαπάνη τουλάχιστον 1 στα 5 ευρώ του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κλιματικές δράσεις. Μας άρεσε πολύ ο τίτλος της έκθεσής σας. Ήδη είναι ενδεικτικός ο τίτλος και του περιεχομένου και μια και ο τίτλος ε, κίνησε το ενδιαφέρον μας, φαντάζομαι εξίσου πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι και η ακόλουθη παρουσίαση και φυσικά και η συζήτηση μετά την εισαγωγή που θα μας κάνει το μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Με την δέουσα προσοχή είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την παρουσίαση της κυρία σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα σας παρουσιάσω την έκθεσή μου με τη βοήθεια κάποιων διαφανειών. Ο Βέτραν Τόγκη ε, είναι ο επικεφαλής ε, για την υπόνηση αυτή, του επιτελείου μου για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης και η Κατρίνα Ντράι που επίσης συνέβαλε τα μάλα στην κατάρτισή της. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Κέστη Κάλου Λάιτ που είναι επίσης συναρμόδια μαζί μου για το, την ειδική αυτή έκθεση πριν να εγκαταλείψει το ελεκτικό συνέδριο για να γίνει πρόεδρος της Εστονίας. Η έκθεση δημοσιεύτηκε στις 22 Νοεμβρίου. Είχαμε μάλιστα πολύ επικοδομητικές συναντήσεις στις 28 Φεβρουαρίου με τον Επίτροπο Αρίας Κανιέτε, τον Επίτροπο Χόγκαν και τον Επίτροπο Μέρδας. Μάλιστα έτυχε θετική υποδοχή ε, στην αρμόδια ομάδα εργασία του Συμβουλίου στι 14 Φεβρουαρίου έκθεση και στην ε, Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού στι 28 Φεβρουαρίου. Εγώ θα σα μιλήσω για την έκθεση, τα πορίσματά τη καθώ και τι συστάσεις τη. Καταρχήν ω προ προς την έκθεση ελέγχου η βασική ερώτηση ήταν το κατά πόσο στόχο τη δαπάνη 1 στα 5 ευρώ της Ευρω... του ενωσιακού προπολογισμού για συναφή με το κλίμα δράση έχει υλοποιηθεί και τι προσθέμενη αξία προσφέρει. Γιατί αν είχαμε 20% δαπάνε, θα είχαμε 212 ε, δισεκατομμύρια δράσεις που θα πρέπει να αφιερώνουμε στην ε, περίοδο προγραμματισμού για, τις... για το περιβάλλον. Μεταξύ του Οκτωβρίου 2015 ε, και το Φεβρουάριο του 2016 κάναμε επισκέψεις ελέγχου στην ε, Πολωνία. Ήμουν μάλιστα παρόν με θέμα την ε, συνοχή και την κοινή γεωργική πολιτική. Στη Γερμανία και τη Ρουμανία για την συνοχή και στην Γαλλία και Ισπανία για την κοινή γεωργική πολιτική. Επίσης είχαμε και έλεγχο για τον ορίζοντα 2020, την Αλία και το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και για όλα αυτά είχαμε πολύ αγαστή συνεργασία. Δεν εξετάσαμε τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον που προκαλούν κάποιες άλλες κοινοτικέ δαπάνες ή μη συναφήσουμε το περιβάλλον ή το κλίμα ενωσιακές δαπάνες. Επίσης, κάποιες άλλες συναφή με το κλίμα δαπάνες εκτός του ευρωπαϊκού προπολογισμού των ε, της επενδυτικής ε, τράπεζας, ας πούμε, δεν ε, καλύφθηκαν από την έκθεση. Ούτε, ούτε αναφερθήκαμε στις πραγματικές δαπάνες, γιατί εδώ μιλούμε για στοχευμένες σχεδιασμένες δαπάνες για την περίοδο 2014-2020. Και ακόμη πραγματικές δαπάνες ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Γι' αυτό μιλήσαμε μόνο για τις προσχεδιασμένες, στοχευμένες δαπάνες. Ποια, τι λένε τα πορίσματα. Φιλόδοξο έργο έχει ξεκινήσει και γενικώ έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό κίνδυνος ανεπάρκειας. Γιατί βρήκαμε καλύτερες και πιο στοχευμένες ε, δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Αλλά στα θέματα της γεωργίας, της ανάπτυξης της υπαίθρου και της αλίας, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεν βρήκαμε σημαντική μεταστροφή προς πιο όφυλο περιβαλλοντικές ε, δράσεις υπέρ του κλίματος. Και η δράση επίσης υστερεί σχετικά του στόχου του 35%. Σε τη φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μερίδιο ε, των περιβαλλοντικών δαπανών ήταν 17,6% μεταξύ 2014 και 2016. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διάμεση αναθεώρηση ε, είπε ότι 18,1% θα δαπανηθεί για τις κλιματικές δράσεις μεταξύ 2014 και 2020. Κάτι που βέβαια πάλι υπολείπεται σε σχέση με τα τουλάχιστον 20% που είναι ο στόχος για τις ε, δαπάνες αυτές. Πάντως αυτά είναι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνουν κατά τη γνώμη μας και κάποια υπερεκτίμηση. Στο δικό μας έλεγχο αναλύσαμε τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επισημάνομαι που κατά τη γνώμη μας δεν ε, ακολουθούσε κάποιες ε, διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Γενικώ, τα πορίσματα στην ε, Γεωργία και την ανάπτυξη Πέθρου ε, εμείς υπολογίσαμε 33 δισεκατομμύρια λιγότερα για κλιματικές δράσεις και οι υποθέσεις που αφορούν τη συμβολή της Γεωργίας και από τις άμεσες ενισχύσεις της γεωργίας ε, δεν ε, συνοδεύονται από ε, κατάλληλες αιτιολογήσεις. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε 20% για άμεσες ενισχύσεις χωρίς, εκτός του πρασινίσματος ως συναφής προς το κλίμα. Αλλά είναι πολύ με, μετριοπαθής η συμβολή στο θέμα της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Επίσης σκέφτηκε να αφιερώσει 10% αντί για 20% η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν η αρχή της συντηρητικότητας που ε, ανέπτυξε η Παγκόσμια Τράπεζα εφαρμοστεί, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η χαμηλότερη εκτίμηση του 10%. Οπότε μειώνεται η συνεισφορά κατά 9 δισεκατομμύρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά πιο ουσιαστικά την ε, ανάπτυξη πέθρου, εκεί είδαμε ε, υπερεκτίμηση κατά 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε μια μεθοδολογία που δεν κάνει επαρκή διάκριση μεταξύ των διαφορών μέτρων. Τώρα, για αντίστοιχα θέματα στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Ταμείο Συνοχής, ε, ένα άλλο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγγιο, εφάρμοσε πιο διεξοδική προσέγγιση. Δεν συνιστούμε λοιπόν μια περιτά γραφειοκρατική, υπερβολικά γραφειοκρατική προσέγγιση. Γενικώ πάντως δεν είδαμε σημαντικές ποιοτικέ αλλαγές στη διαχείριση των δαπανών της κοινή γεωρικής πολιτικής, ιδιαίτερα για σημαντικά οικονομικά μέτρα. Αλλά ε, είδαμε κάποια παραδείγματα καλύτερης στόχευσης και των πρακτικών. Για παράδειγμα, στο σχεδιασμό κάποιων δασοκομικών μέτρων και στις τρεις περιφέρειες που επισκεφθήκαμε, για την αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, για παράδειγμα, ή για το σχεδιασμό αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων. Στην Ανδαλουσία, για παράδειγμα, όπου η διάβρωση του εδάφους ε, παρεμποδίζει την ανάπτυξη της ε, παραγωγής ελαιοδέντρων. Επίσης, ε, στη Γαλλία είχαμε την το παράδειγμα ε, παραγωγής ενέργειας από απόβλητα. Τα μισά είναι γεωργικά απόβλητα και τα άλλα πράσινα απόβλητα. Υπάρχει α, ε, χρόνος ακόμη για αλλαγές στην παρούσα περίοδο προγραμματισμού και ποιοτικά και ποσοτικά. Η Γενική Διεύθυνση θα μπορούσε να αυξήσει τον εξορθολογισμό της α, ε, κλιματικής δράσης με νέα στοχευμένα μέτρα και να χρησιμοποιήσει την ενδιάμεση αξιολόγηση για να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020 και επίση θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και τις διαβουλεύσεις για το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής που πρόσφατα ξεκίνησαν από τον Επίτροπο Χόγκαν για να γίνει καλύτερος προγραμματισμός του μέλλοντος της Επιτροπής Γεωργίας. Πάντως η γεωργία και η ανάπτυξη πέθρου δεν θα είναι οι μόνοι τομεί ε, στους οποίους μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα για τις κλιματικές αλλαγές. Στην έρευνα, το ορίζοντας 2020 επίσης υπολείπεται του στόχου του 35%. Θα αντίθεση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής είχαμε μία μεταστροφή προ περισσότερε φιλοπεριβαλλοντικέ δράσει και είχαμε αύξηση από 12% στην προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο σε 21% στην παρούσα χρηματοδοτική περίοδο. Και επίσης καλύτερη στόχευση, καλύτερη εστίαση στη Γερμανία, Πολωνία και Ρουμανία για παράδειγμα είδαμε περισσότερες δαπάνες για μέτρα που έχουν 100% περιβαλλοντική εστίαση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όμως τα προγράμματα που έχουν προσημειωθεί για περιβαλλοντικές δράσεις ε, είναι μόνο 1,4% των 83 δισεκατομμυρίων ε, ευρώ που είναι διαθέσιμα. Ε, καταλήξαμε λοιπόν σε 7 συμπεράσματα που θα τα συνοψίσω αναφέρονται σε αυτή τη διαφάνεια. Καταρχήν θέλουμε μία ε, στιβαρή ετήσια ε, προσπάθεια εξυγίανσης, ε, ένα πλαίσιο περιεκτικό για την υποβολή εκθέσεων, αρχική αξιολόγηση, εκτίμηση των περιβαλλοντικών αναγκών ή των κλιματικών αλλαγών, ιδιαίτερα με βάση τις παγκόσμιες εξελίξεις, ώστε να διορθωθούν οι υπερεκτιμήσεις που εντοπίστηκαν στην έκθεση. Επίσης, ε, να γίνουν ε, σχέδια δράσης για τις περιοχές που υστερούν και τους κανόνες που, και τους τομείς που υστερούν και να γίνει έλεγχος των πραγματικών δαπανών και των πραγματικών αποτελεσμάτων. Και τέλος, διερεύνηση όλων των πιθανών δυνατοτήτων, ώστε να έχουμε μια ουσιαστική μεταστροφή προς πραγματικές κλιματικές δράσεις. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κύριε Όεν. Περνάμε στη συζήτηση. Πρώτος ε, ζήτησε το λόγο ο κύριος Άγνιου. Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το θέμα το έχω ανιστερνιστεί και βλέπω από την έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να δαπανίσει 36 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να βελτιώσει τον κόσμο, είτε μειώνοντας τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με άλλα μέτρα. Τεράστιο το ποσό αυτό. Εν τω μεταξύ όμως επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε υποδομέ, μεταφορέ, φορτηγά, αεροπλάνα χρησιμοποιούνται όλα αυτά, άρα δηλαδή ε, από αυτά και μόνο, επειδή θα παράγουν διοξείδιο το άνθρακα, αυτό είναι αντιφατικό. Ε, δεν χρειάζεται να δαπακανά κανεί χρήματα για να πει στου ανθρώπου ότι δεν πρέπει να ασχολούνται με τη χειρουργία ή πρέπει να σταματήσουν να ταξιδεύουν. Αν πιστεύει κανεί ότι πρέπει να μειωθούν οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, ε, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πει στου ανθρώπου να μην κάνουν τίποτα, να παραμένουν αδρανεί. οι Ανατολικογερμανοί λένε ότι ίσως κάποιος ασβεστόλιτος ε, να μην είναι καλός, ε, θέλουν να τον μεταφέρουν από αλλού, από πολύ μακριά. Ε, και Γι' αυτό πρέπει να γίνονται οι μεταφορές. Όμως αυτό καθιστά την ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο δαπαναλή. Το ίδιο ισχύει και για τις καλλιέργειες. Αναφέρεται η δασοκομεία, αλλά δεν είναι το αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχω πει πανελειμμένα, πολλοί θεωρούν ότι η δασοκομεία παραμένει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως κάτι όπου μπορούμε να δαπανίσουμε χρήματα και αυτό είναι άμεση επίπτωση και παρενέργεια του κλίματος κλίματος έχουμε έντονες βροχοπτώσεις ε, κατά καιρού ε, και ακούμε ότι ε, γίνονται κατασκευές σε περιοχές που δεν θα έπρεπε. Πού καταλήγουν όλα αυτά? Στις πλημμύρες. Δεν είναι ότι βρέχει περισσότερο, απλά προκαλούνται ζημιές λόγω των αιτιών που σας ανέφερα. Μπορεί λοιπόν κανείς να δαπανίσει χρήματα για να ε, μπορέσει να μεταφαρμόσει άλλα μέτρα τα οποία θα παρεμποδίσουν τις ζημιές ε, από την κλιματική αλλαγή. Δεν γίνεται όμως λόγος για αυτά στην έκθεση. Κάτι άλλο που νομίζω το αναφέρει η έκθεση είναι ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στο στόχο να δαπανώνται 30 δις το χρόνο ε, για την ε, γεωργία και από την άλλη να περιστούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πώς μπορείτε να αποδείξετε ότι τελικά αυτή η δαπάνη των 30 δις θα είναι αιτιολογημένη και θα δαπανηθούν σωστά τα χρήματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Άγνιου. Άλλος κανείς παρακαλώ. Ο κύριος Χόισλεγκ. Θέλω να πω ότι ο κύριος Αγνιού δεν είναι ο μόνος ε, που ήθελε να τοποθετηθεί στην έκθεση. Εγώ το βρίσκω περίεργο το ότι ένα κόμμα που θέλει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να σκέφτεται ε, το τι θα κάνουμε εμείς στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κοιτάξτε λιγάκι τη δική στη δουλειά, να μην ασχολείστε με τα δικά μας, ε, δεν χρειάζεται. Σιγά σιγά και με ασφάλεια μπορείτε να βγείτε στη σύνταξη, να μην ασχολείστε τα δικά μας τα θέματα, γιατί για το κλίμα, σκύλος εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Αν όμως δει κανεί τα διάφορα μέτρα τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να συγκεντρώσουμε, θέλω να πω το εξή. Ε, ε, τα χρήματα δαπανώνται κάπως αντιφατικά τα κονδύλια. Ε, προηγουμένως αναφερθήκατε στο βιοαέριο. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν θέλουμε να παράγουμε ενέργεια από τη γεωργία, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση καταλήπων και όχι όπως ε, λανθασμένα ε, έχει γίνει στη Γερμανία με την καλλιέργεια ραβοσίτου και μονάδες παραγωγής ε, βιοαερίου. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Να χρησιμοποιούμε τα απόβλητα και τα κατάλοιπα και έτσι να παράγουμε ενέργεια από τη γεωργία. Γιατί αυτό που πιστεύαμε πολύ μας παλαιότερα, ότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό, δεν υπάρχει αυτό. Ε, πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή την άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό παραγωγής ενέργειας ε, από τη Γεωργία. Πρέπει λοιπόν να ε, απελευθερωθούμε από αυταπάτες. Ε, είχαμε και τη συζήτηση για το φινικέλαιο, ότι το φινικέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενέργεια, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι αντιπαραγωγικό το φινικέλαιο για την παραγωγή ενέργειας. Ως εκ τούτου, αυτά που γίνονται κάτω από την ε, προστασία του κλίματος ε, θα πρέπει να τα εξετάσουμε ενδελεχέστερα. Και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να εξετάσουμε κυρίως τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα, κατά πόσο τα μέτρα αυτά πραγματικά εξυπηρετούν το στόχο προστασίας του κλίματος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για όλα αυτά που είπατε. Ε, πολύ συγκεκριμένα για το σημείο υπερθμών 7 στην έκθεση. Έχω μία ερώτηση. Αν είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα πρόγραμμα δράσης και υπάρξει τελικά αυτό το πρόγραμμα, εμένα με ενδιαφέρει ποια είναι τα τρία σημεία τα οποία κατά την άποψή σας είναι τα σημαντικότερα στον τομέα της γεωργίας. Να μας πείτε λιγάκι ε, τι είδου σκέψεις έχετε, εκφράστε μας ε, τις σκέψεις σας, γιατί αυτό ίσως να μας έδινε και μας μια ιδέα προς τα που βαδίζει το τρένο. Ε, και άλλη μια ερώτηση για το σημείο υπαριθμών 10. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε εσεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση, και αυτό δεν το λέω ειρωνικά, αλλά πραγματικά, πώ πιστεύετε ότι η Κομισιόν είναι σε θέση να ε, αποφανθεί τον όγκο των κονδυλίων που είναι απαραίτητα για την προστασία του κλίματος. Υπάρχει έτσι μια τάξη μεγέθους ή είναι εμβαλωματικές αυτές οι απόψεις για διάφορους τομείς. Ο τρίτος τομέας αφορά τις ε, άμεσες ενισχύσεις στη Γεωργία. Ε, πιστεύετε ότι με τις ε, άμεσες ενισχύσεις μπορούμε να περάσουμε σε μια αλλαγή, δηλαδή να καταβάλουμε ενισχύσεις και με βάση την προστασία του κλίματος και θεωρείτε ότι με το 20% αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε, αν τολμήσουμε βέβαια. Κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ αυτούς που προετοίμασαν την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να μου πείτε, καταρχήν, οι άμεσες αυτές πληρωμές δεν απευθύνονται για θέματα αλλαγής κλίματος. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε λοιπόν ποια είναι η θέση σας όσον αφορά το θέμα αυτών των άμεσων ε, επιδοτήσεων. Τώρα, όσον αφορά την ε, λέξη που χρησιμοποιήσετε εδώ, τι είναι ακριβώς αυτή η φιλική προς το περιβάλλον και προς την αλλαγή του κλίματος, Γεωργία. Τρίτον, υπάρχουν πολλά που γίνονται στα κράτη-μέλη και για να μην είμαστε άδικοι στις ε, επικρίσεις μας, Κοιτάξτε παραδείγματο χάρη το θέμα των εκπομπών, το θέμα της κτηνοτροφίας, ε, ιδιαίτερα για τα βοηδή. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες ε, για τις μετρήσεις αυτών των εκπομπών και για να υπάρχει μια γεωργία και μια κτηνοτροφία λίγο πιο φιλική προς το περιβάλλον και Νομίζω ότι η κριτική σας είναι πολύ αυστηρή. Δεν είστε πολύ δίκαιοι όσον αφορά αυτά που έχουν γίνει. Για σας τι είναι μια πιο αποτελεσματική γεωργία. Ίσως εδώ μπορούμε να αλλάξουμε και τους όρους που χρησιμοποιούμε, την ορολογία. Διότι πολλοί γεωργοί προσπαθούν και πολλοί κτηνοτρόφοι προσπαθούν να είναι πιο αποτελεσματικοί και να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Συγκεκριμένα λοιπόν, τι θα προτείνατε εσείς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω για την ε, παρουσίασή σας. Πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί πολύ. Σίγουρα η δράση μας για να εκπληρώσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει που είναι στόχοι συνολικοί βεβαίως, δεν αφορούν μόνο τη γεωργία, θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μία πιο ολοκληρωμένη δράση. Βεβαίως αυτό έχει ένα κόστος και σήμερα γνωρίζουμε ότι στην ενιαία αγορά υπάρχουν πολλές διαφορετικές, παραδείγματο χάρη μεταξύ του Βορρά και του Νότου της Ευρώπης ή της Ανατολής και της Δύσης θα ήθελα να μου πείτε η στήριξη που μπορούμε να δώσουμε στους γεωργούς, η οποία σήμερα διαφέρει. Οι άμεσες πληρωμές, παραδείγματο χάρη, πολλές φορές είναι το πενταπλάσιο σε κάποιες περιοχές αυτών που είναι αλλού. Παρ' αυτά, όλοι οι γεωργοί, όπου και αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν να τηρήσουν τα ίδια ε, αντικειμενικά κριτήρια και έχουν να υλοποιήσουν τους ίδιους στόχους. Για κάποιους λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι για άλλους. Είναι πολύ πιο δύσκολο να συμμορφωθεί κανείς με όλα αυτά τα προαπαιτούμενα, καθότι χρειάζονται επενδύσεις παραδείγματο χάρη. Χρειάζονται επενδύσεις ε, πέρα από τις άμεσες πληρωμές και πολλές φορές βλέπουμε ότι οι τιμές αγοράς των προϊόντων στην Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερες ε, σε σχέση με αυτές ε, στις δυτικές χώρες Ευρώπης. Η δράση λοιπόν για την προστασία του περιβάλλοντος και η δράση που αφορά την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να βασίζεται σε ένα πιο δίκαιο σύστημα, σε πιο δίκαια κριτήρια. Κατά την άποψή σας θα πρέπει να λειτουργήσουμε αποκεντρωμένα Μήπως πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ο πυλώνας, ο δεύτερος πυλώνας και οι δυνατότητές τους. Γιατί βλέπουμε σήμερα να υπάρχουν πολλές διαφορετικές αρχές που μπορεί να ορίσουν τις δραστηριότητες που θα επιλεγούν. Και αυτό άσχετα με τη στήριξη που θα λάβει ο κάθε γεωργός. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω Πρόσεξα ότι η ανάπτυξη της Υπέτρου και οι πληρωμές ε, που αφορούν την ανάπτυξη της Υπέτρου έχουν μειωθεί κατά 2 με 3% τα τελευταία χρόνια. Ενώ είναι σαφές ότι αυξάνονται τα ποσά που διατίθενται για την ε, αλλαγή του κλίματος και τις δράσεις που αφορούν την αλληλεγγύη. Πώς μπορούν λοιπόν οι γεωργοί να υλοποιήσουν όλα αυτά που αφορούν το κλίμα, ενώ την ίδια ώρα βλέπουμε ότι οι αγορές έχουν υποστεί σημαντικές πιέσεις για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα στον τομέα του ίνου, παραδείγματος χάρη, στα οπροκυπευτικά. Θα πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές όταν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψετε να επανέλθω κύριε Πρόεδρε και έπρεπε να το κάνω γιατί ε, αναφέρθηκε κάτι επί προσωπικό, αναφέρθηκε το όνομά μου και κάποιος είπε γιατί θα πρέπει να ανησυχώ γιατί θα έχουμε το Brexit, θα φύγει η Μεγάλη Βρετανία. Ο λόγος που ανησυχώ είναι ο εξή, γιατί μιλάμε για 30 δις ευρώ σε αιτήσια βάση για να βελτιωθεί ο καιρό ε, στον κόσμο και ε, όμως ένα μεγάλο ποσό θα το συμβάλλουν οι Ευρωπαίοι, ε, με συγχωρείτε, οι Βρετανοί φορολογούμενοι. Εγώ τους εκπροσωπώ. Και παρέχουμε σε αυτό που έχει ελεγχθεί ως σύνθημα «No taxation without representation». Να μην επιβάλλονται φόροι αν δεν υπάρχει και η σωστή εκπροσώπηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης ε, και για την έκθεση που ακούσαμε σήμερα. Οι συνάδελφοί μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι και εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός ε, όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος ε, που οφείλεται σε ανθρώπινες παρεμβάσεις. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε γιατί είχαμε παλαιότερα κατά τον Μεσαίωνα εποχές όπου στα μοναστήρια βλέπαμε τελείως διαφορετικά λουλούδια. Αυτά το 1000, 1200 και μέχρι σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να εγκρίνει αυτό το ποσό ότι χρειαζόμαστε 30 δις για τη βελτίωση του κλίματος. Εσείς το λέτε αυτό, ενώ εχθές είδαμε μια έκθεση όπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών λόγω του λοιμού στην Ανατολική Αφρική διαμαρτυρήθηκε ότι ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να διαθέσει 4 μόνο δισεκατομμύρια ευρώ για να σωθούν άνθρωποι, να σωθούν 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ το βρίσκω ανεύθυνο. Ανεύθυνο το ότι θέλουμε να κάψουμε στην κυριολεξία 30 δις και αυτά τα 4 δις για την Ανατολική Αφρική λέμε ότι δεν τα έχουμε. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλον κανένα να θέλει το λόγο από την Ομίγυρη. Οπότε θα παρακαλέσω τον καλεσμένο μας από το Ενεκτικό Συνέδριο να λάβει το λόγο για να δώσει απαντήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και όλα τα μέλη που έθεσαν ε, ερωτήσεις. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά και με μεγάλη χαρά άκουσα όλες τις ερωτήσεις Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, ξεκινώντας ε, από την ερώτηση του κύριου Άγνιου που έγινε και πρώτη. Μάλιστα θα απαντήσω από κοινού με την τελευταία ερώτηση του κυρίου Ντές. Είπατε κύριε Άγνιου ότι είμαστε διατεθειμένοι να δαπανίσουμε 300, 30 ε, εκατομμύρια για να βελτιώσουμε τον καιρό. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο. Κανένα κονδύλιο δεν προτίθεται να αλλάξει τον καιρό. Και Μιλήσατε για την ε, σημασία να κοιτάξουμε και το υπόλοιπο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όλες αυτές τις δαπάνες, παραδείγματο χάρη στις υπεδομές, τις μεταφορές. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό τα ποσά τα οποία έχουν περάσει από τον ε, λογιστικό έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν έχουμε ακόμα ελέγξει αυτές τις δαπάνες που αφορούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός αυτών που στοχεύουν το κλίμα. Και βεβαίως πρόκειται για ποσά που φτάνουν και το 80% αυτού του τομέα. Μπορείτε να κοιτάξετε στον ιστότοπο του ελεγκτικού συνεδρίου μία σειρά εκθέσεων, όπως αυτή εξάλλου που παρουσίασα σήμερα, πριν από δύο χρόνια παραδείγματο χάρη, δημοσιεύσαμε μια έκθεση για τα περιφερειακά αεροδρόμια και την ε, ε, μελέτη σκοπιμότητας που έγινε για αυτά. Εκεί μπορείτε να δείτε ακριβώς για την περίοδο μετά το 2008, περιοχή ύφεσης, περίοδο ύφεσης, και την χρήση αυτών των περιφερειακών αερολιμένων και αν πραγματικά αξίζει η επένδυση είναι ένα είδος απάντησης ε, στην ε, ερώτησή σας. Κοιτάξτε αυτή την έκθεση, αφορά υποδομές στον τομέα των μεταφορών. Καταλαβαίνετε όμως ότι και το θέμα των μεταφορών αφορά την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Είναι μια άλλη πτυχή απλώς αυτής της ε, ανάλυσης. Είπατε ότι κατά την άποψή σας ένα σοβαρό πρόβλημα είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες και βεβαίως ε, η ανθρώπινη δράση και παρέμβαση. Εάν σας ενδιαφέρει αυτό, εμείς σαν ένας ανεξάρτητο οργανισμός, το ελεκτικό συνέδριο, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της πλημμύρας που βεβαίως έχει πλήξει πάρα πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι είναι συναφές το θέμα αυτό με την αλλαγή του κλίματος. Εγώ μάλιστα θα θα εργαστώ μαζί με τον συνάδελφο που βρίσκεται στα αριστερά μου για το θέμα αυτής ακριβώς ε, της ε, έκθεσης ε, με θέμα τις πλημμύρες. Και θα δημοσιευθεί μάλιστα το 2018 η έκθεση αυτή. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα που θίξατε, δηλαδή τις συνέπειες των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τι επιπτώσει, τη εκπομπέ, διοξιδίου του άνθρωπου. Έχετε δίκιο. Έχει εξεταστεί το θέμα αυτό πολύ παλιότερα και βεβαίω αυτό αφορά τον συνολικό προπολογισμό στο μέλλον. Σίγουρα θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει όχι τις προβλεπόμενες δαπάνες, αλλά τις πραγματικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας δείκτες που να αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Και έχετε δίκιο που πήγεται αυτό το θέμα. Νομίζω, κύριε Ντές, αυτό απαντά και στην δική σας ερώτηση. Δεν θέλω τώρα να μπω στην ε, μεγάλη συζήτηση για το αν ναι ή όχι υπάρχει αλλαγή του κλίματος. Ε, εδώ συζητούμε για τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος ε, επί της γεωργίας. Το θέμα της ανθρωπογενούς ή όχι αλλαγής του κλίματος και ποια είναι η ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτό. Η αύξηση της θερμοκρασίας από το 1951 μέχρι το 2010 και αν αυτό οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες, αν είναι ανθρωπογενής, αν η αύξηση των εκπομπών του ε, προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Νομίζω ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν επιστήμενες που πρεσβεύουν οι περισσότεροι αυτήν την θεωρία και άλλοι όχι. Αναφερθήκατε στα θέματα των, ε, της ε, βιομάζας, της χρήσης ε, κάποιων καλλιεργιών. Φέρετε και μάλιστα το παράδειγμα του Καλαμποκιού στη Γερμανία για τη δημιουργία βιομάζας και αυτό είναι κάτι που βεβαίως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην η υπόσχεση του 25% του προϋπολογισμού που θα πρέπει να διατεθεί για αυτές τις δράσεις, ένα ευρώ στα 5. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή, αν θέλετε, υπόσχεση. Και θα πρέπει να δούμε πώς ε, οι επαληθεύσεις, πώς η παρακολούθηση ε, των εκπομπών, παραδείγματο χάρη, θα γίνει με πιο σοβαρό τρόπο και όχι μόνο τις δαπάνες που μέχρι τώρα είναι αφιερωμένες στην δράση αυτή. Και αυτό βεβαίως θα αποτελέσει και το αντικείμενο της άλλης έκθεσης που θα δημοσιευθεί αργότερα το καλοκαίρι. Αναγνωρίζω βέβαια κάποια από αυτά που είπατε όσον αφορά τον τρόπο μέτρησης στο παρελθόν και κοιτάξτε την έκθεσή μας ε, στην ιστοσελίδα μας ε, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από ένα χρόνο. Κυρία Νίλ. Κυρία Νόιφελ. Η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η ανάπτυξη πέθρου σίγουρα μπορεί να γίνει με πολύ καλύτερο τρόπο και μάλιστα ακούσατε και τον Μόδιο Επίτροπο πολύ πρόσφατα. Είναι όμως, αν θέλετε, ίσως αργά για νέο σχέδιο δράσης το σημερινό πολιετές ε, ε, σχέδιο. Η ομάδα του Καρλ Μέρντες Η ομάδα του Επιτρόπου Μουέντας, έτσι και αλλιώ έχει υποβάλει κάποιες προτάσεις. Η ιδέα μας είναι να συνεχιστεί το σχέδιο δράσης, εντοπίζοντας στην έκθεσή μας κάποιους τομείς που σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική η δράση μας. Αλλά και η Επιτροπή και το Συμβούλιο και εσείς σαν νομοθετικές αρχές μπορείτε να υποβάλλετε ε, τις δικές σας προτάσεις. Ε, μιλήσατε έτσι κι αλλιώς ε, και για την άλλη έκθεση που αφορά τις επιπτώσεις επί της γεωργίας της δράσης για το περιβάλλον, αλλά και η δική μας έκθεση εμπεριέχει κάποιες προτάσεις, όπως παραδείγματο χάρη καλύτερη κατάρτιση για τους γεωργούς, ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στον τομέα αυτό για μια πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική δράση. Το θέμα της ε, γεωργίας και των πληρωμών που θα πρέπει να εξαρτώνται από την δράση και το περιβάλλον, περισσότερο τουλάχιστον να εξαρτώνται από αυτή τη δράση στο μέλλον. Νομίζω ότι και εδώ πρέπει να ακούσουμε τον Επίτροπο Χόγκαν, ο οποίος με πολύ ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι θα πρέπει και η γεωργία και όλος ο τομέας της γεωργίας να συνεισφέρει πολύ περισσότερο στη γενικότερη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και την αλλαγή του κλίματος. Νομίζω ότι ε, αυτές είναι οι οδηγίες που ο Φιλ Χόγκαν έδωσε προς την ομάδα του, προς τους συνεργάτες του και σίγουρα η δική μας ε, μελέτη, καθώς και η μελέτη για το πρασίνισμα που θα δημοσιευθεί αργότερα, το 2017, σίγουρα μπορεί να αποτελέσει βάση για κάποιες ε, προτάσεις. Κυρία Μαγκίνες, νομίζω ότι είδατε κάπως ε, αρνητικά αυτά που δημοσιεύσαμε δεν είμαστε τόσο αρνητικοί. Αν κοιτάξετε και την ετήσια έκθεση για τη συμμόρφωση θα δείτε ότι δεν είναι τόσο αρνητικά τα σχολεία μας. Εδώ πρόκειται για μία έκθεση που προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε σας έδειξα μάλιστα και κάποιες πολύ, συγκεκριμένα παραδείγματα για την ενέργεια, για την αποτελεσματικότητα και την απόδοση την ενεργειακή. Έδωσα κάποια πολύ θετικά παραδείγματα στο Παρίσι, στο Βουκουρέστι. Κάποιες ε, δαπάνες συνοχής δεν ε, είναι μόνο αρνητικά τα σχόλιά μας. Προσπαθήσαμε να είμαστε πιο ισορροπημένοι στην παρουσίαση που κάναμε. Επίσης παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ε, αναδάσωσης. Θελήσαμε παρόλα αυτά να εντοπίσουμε τους τομείς αυτούς όπου υπήρξαν και κάποιες ε, υπερεκτιμήσεις και στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. 9 και 24 δις. Ε, εκεί σαφώς και υπάρχουν υπερεκτιμήσεις, παρουσιάζουμε τους αριθμούς. Κύριε Ρόπε, λέτε ότι δεν είναι εύκολο να συμμορφωθούν οι γεωργοί, ότι είναι περίπλοκο το σύστημα, το ελεγκτικό συνέδριο και στην ε, ετήσια έκθεση, αλλά και σε αυτήν την ειδική έκθεση. Και εδώ και χρόνια μάλιστα αναφέρουμε το πόσο περίπλοκο είναι το σύστημα και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί λέγοντας ότι σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η περιπλοκότητα δεν είναι κάτι που βοηθάει τους ε, Ευρωπαίους σε όλους τους τομείς να συμμορφωθούν. Βέβαια δεν είναι εύκολο να υπάρξει και η απλοποίηση. Έγινε μια καλή αρχή από τον Επίτροπο. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει όλα να πεταχτούν στα σκουπίδια. Λέμε ότι οι βελτιώσεις θα πρέπει να συνεχιστούν, θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες. Και όσον αφορά την ε, δράση για την αλλαγή του κλίματος, Σίγουρα οι δαπάνες όταν αποφασίζονται και όταν ε, ψηφίζονται θα πρέπει να εμπεριέχουν και μια συνιστόσα που να αφορά άμεσα την αλλαγή του κλίματος. Και βεβαίως και είναι περίπλοκο το σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, αλλά σίγουρα χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια για να γίνει πιο σαφές και πιο απλό το σύστημα. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Could I add one other thing? Θα μπορούσα να προσθέσω κάτι ακόμη και ευχαριστώ θερμά την γραμματεία που μου την υπενθύμησε. αν σας βοηθά αυτή η ειδική έκθεση και η σημερινή συζήτηση, ε, το πρώτο τμήμα του ελεκτικού συνεδρίου, στο οποίο εγώ είμαι αρμόδιος ε, για τη βιώσιμη χρήση των ε, φυσικών πόρων, θα εκπονήσει και άλλες ειδικέ εκθέσεις που έχουν κάποια συνάφεια με το έργο της Επιτροπής σας. Πέντε νέες εκθέσεις έχουν προγραμματιστεί για φέτος Ξέρω ότι είστε πολύ απασχολημένοι και ίσω ε, δεν θα προλάβετε να τι εξετάσετε όλε. Πάντω, οι πέντε είναι οι εξή. Ένα αφορά του φορεί πιστοποίηση για τον έλεγχο των δαπανών. Θα δημοσιευθεί το Μάιο. Έχουμε μια άλλη έκθεση ειδική για τους νέου γεωργούς που θα δημοσιευθεί Ιούνιο με Ιούλιο φέτος. Μια άλλη έκθεση για το, το προγραμματισμό τη αγροτική ανάπτυξη στι αρχέ του Οκτωβρίου. Ένα για το σύστημα βασικών πληρωμών που αναμένεται για τα τέλη του Οκτωβρίου τρέχοντος έτους και ένα που ανέφερε και ίσως είναι και πιο ενδιαφέρουσα για σας θα αφορά το πρασίνισμα, greening, και θα δημοσιευθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Και στο ελεκτικό συνέδριο έχουμε διάφορα μέλη που είναι επιφορτισμένα με διαφορετικά θέματα. Ίσως ε, θα σας ενδιαφέρει και το θέμα για την ενέργεια και το κλίμα, η σχετική δημοσία έκθεση για την οποία επίσημα αρμόδιος εγώ. Οπότε, εκτός από αυτές τις έξι δικές εκθέσεις, ε, ίσως χρειαστεί να προσκαλέσετε και άλλα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου για να σας εξηγήσουν το έργο μας, γιατί προσπαθούμε να είμαστε ανεξάρτητοι, αντικειμενικοί, αμερόληπτοι και να εγκύπτουμε μόνο στα στοιχεία. Ε, σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Μήπως ε, θέλει κανείς το λόγο για επερώτηση. Κυρία Μαγκίνες. Σας ευχαριστώ που μας προαναγγείλατε κάποιε μελλοντικέ εκθέσει. Μερικέ όντω ε, μα ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, εμένα με ενδιαφέρει αυτή για του νέου γεωργού, γιατί θα κάνει μια ανάλυση των μέχρι τώρα μέτρων τη ε, μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ και θα κάνει και έναν απολογισμό των μέτρων αυτών για να δούμε τι πήγε καλά και τι στραβά. Ε, Επίση, ε, χαίρομαι που ε, <laughs> σας ενέπνευσε αυτή η πασχαλινή περίοδος και υπάρχει μια μεγαλύτερη ε, μια πιο ευδιάθετη κατάσταση και πρόσθεσε και ο κύριος Άγγινος αυτά το δικό του χαμόγελο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Και σας κύριε Βουίν και τους συνεργάτες σας. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο το έργο σας και πολύ πλούσια η εμπειρία του ελεκτικού συνεδρίου και πολύ διεξοδικές οι αναλύσεις που πραγματοποιεί. Σας ευχαριστούμε και πάλι και εμείς θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Τακτικά έχουμε ενημέρωση από τους συγγητές μας για την πορεία των εκθέσεών τους και την πορεία των τριμερών διαλόγων. Μας ενημερώνουν ε, για την πορεία των τριμερών διαλόγων, ε, τις εκκρεμότητες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αυτά τα εξετάζουμε και στους συντονιστές. Θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Μάρτιν Χόισλινγκ την ενημέρωση για τους τρέχοντες τριμερείς διαλόγου για τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Μα Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ ε, που μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, ε, γιατί έχω την εντύπωση ότι προχωράμε τώρα σε μια τελική φάση. Τελευταία φορά σας είχα πει ότι οι δύο πρώτοι ε, τριμερείς διάλογοι με την Μαλτέζικη Προεδρία δεν ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικοί. Είχαμε την εντύπωση ότι η Μαλτέζικη Προεδρία επιμένει στην εντολή του Συμβουλίου και δεν ενδιαφέρεται να κάνει καμία αλλαγή. Ε, νομίζω ε, καταστήσαμε σαφέ ε, ως διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου ότι πρόκειται για τριμερή διάλογο γιατί όλοι πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς και έτσι κι αλλιώς η Προεδρία του Συμβουλίου πήρε τέτοια εντολή για πρώτη φορά από το Συμβούλιο. Μετά λοιπόν από διμερείς ε, συζητήσεις και όπου ο Επίτροπος ε, είπε ότι θα πρέπει σύντομα να έχει το αποτέλεσμα, αποφασίσαμε να αλλάξουμε τις μεθόδους εργασίας. Υπήρξαν πάρα πολλές ε, συναντήσεις, έτσι ώστε οι συμβαστικές προτάσεις που είναι απαραίτητες για τους τριμερείς διολόγους να καταστεί δυνατόν να προετοιμαστούν. Υπάρχουν ε, ως εκ τούτου τέσσερα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε και ελπίζω να έχουμε πλησιάσει στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πρόκειται καταρχήν για, την, ε, για τα θερμοκήπια από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταθέσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση και ελπίζω να έχουμε και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, η εξαίρεση περιορίζεται σε έξι βόρειες χώρες όπου υπάρχουν ειδικέ συνθήκες και αυτό το ε, συνάγουμε από την οδηγία για τα ε, φυτοφάρμακα, οι χώρες Βαλτική, η Σουηδία και η Δανία. Αυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως εξαίρεση και θα μπορούν να λειτουργούν λειτουργούν διαφορετικά από την Ευρώπη. Το που μας απασχολεί είναι ποιο είναι το ποσοστό το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί από από πλευρά εδάφους και από την ίδια την επιχείρηση. Νομίζω ότι από αυτού ε, θα βρούμε κάποια λύση, ε, θα ικανοποιηθούν οι βόρειε χώρε, ε, θα ληφθούν υπόψη οι κλιματικές ιδιαιτερότητε αυτών των κρατών και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Πλησιάζουμε και στο θέμα της εκπνοής των ρυθμίσεων κατεξαίρεση. Και εκεί πλησιάζουμε σε μια συγκεκριμένη λύση. Το Συμβούλιο φοβάται ότι αν τελικά αυτή την εκπνοή την συνδέσουμε με τράπεζα δεδομένων, αυτό θα δημιουργήσει νέα γραφειοκρατία. Όμως ξέρετε κάτι, τα χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα, γιατί ο ε, καλλιεργητής, ο καλλιεργητής θα πρέπει να ξέρει πότε πρέπει να χρησιμοποιήσει τους οικολογικούς του σπόρους. Αυτό είναι σημαντικό ε, για όσους ασχολούνται με οικολογικές καλλιέργειες. Και εντωμεταξύ νομίζω και το Συμβούλιο κατάλαβε ότι πρέπει να βρούμε ε, μία λύση από αυτού. Για να εκφραστούμε σωστά μπορούμε να πούμε ότι οι εξαιρέσεις ε, εκπνέουν το 2025 ε, και να δώσουμε τη δυνατότητα στους βιοκαλλιεργητές να να παρουσιάσουν ότι πράγματι υπάρχουν αίτια που πρέπει να έχουν εξαιρέσει. Τώρα, όσον αφορά τις τράπεζες δεδομένων για οικολογικά ζώα, bio-animals, ε, τα βιολογικά ζώα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για αυτά σε τράπεζες δεδομένων έτσι ώστε όσον αφορά την εκτροφή αυτών των ζώων με οικολογικές προδιαγραφές πάρουμε τα κοτόπουλα. Κάποιες χώρες έχουν βιολογικά κοτόπουλα, άλλες χώρες πάλι όχι. Η βιολογική εκτινοτροφία λοιπόν ε, μπορεί να κρυθεί κάτω από αυτούς τους όρους. Κατόπιν, όσον αφορά τους σπόρους, ως κοινοβούλιο είπαμε ότι χρειαζόμαστε ειδικές ρυθμίσεις ε, για τους σπόρους και τη σπορά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε η Κομισιόν να καταθέσει νέα πρόταση, ένα νέο κανονισμό για τους ε, σπόρους. Στον οικολογικό τομέα θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να προχωρήσει με τους δικούς του τους ε, σπόρους. Ε, και δεν είναι αλήθεια ότι όλοι οι οικολογικοί σπόροι εντάσσονται στο μοντέλο της παραδοσιακής εκτροφής. Η Κομισιόν έχει κάποια προβλήματα από αυτού και νομίζω τώρα η Κομισιόν υπενήχθη ότι ε, θα υπάρξει κάποια δήλωση προθέσεων. Αλλά ακόμα αυτό δεν είναι σίγουρο. Δεν αποκλείεται βέβαια. Εμείς ε, θέλουμε να ακολουθηθεί η σωστή κατεύθυνση όσον αφορά το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε συνεχώς να το αναβάλουμε το λέμα και να πούμε ότι οι σπόροι, περιμένετε λιγάκι, θα υπάρξει μια νέα ε, ρύθμιση, νομοθετική ρύθμιση και θα ρυθμιστείτε κι εσείς. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα, ένα από τα πιο λεπτά πολιτικά θέματα είναι οι νέες οριακές τιμές για, ε, για τον οικολογικό τομέα. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα οι απόψεις δεν έχουν αλλάξει. Νομίζω ότι στις ε, άτυπες ε, συναντήσεις πλησιάζουν οι περισσότεροι στην πρόταση του Κοινοβουλίου. Η θέση είναι ότι θα περιμένουμε να δούμε την πρόταση της Κομισιόν, να δούμε από πού προέρχονται παραδείγματος οι προσμίξεις. Οι προσμίξεις ε, τι έκταση καταλαμβάνουν. Ε, αφορούν τον παραγωγό, αφορούν τον έμπορο. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτή τη βάση ε, θα μπορέσουμε αργότερα να ξανασυζητήσουμε, γιατί μέχρι τώρα βρισκόμαστε στο σκοτάδι οι βιοκαλλιεργητές λένε ότι εμείς ε, δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό για να καταλήξουμε σε μια ρεαλιστική λύση. Και θέλω να δείξω και ένα τελευταίο θέμα, το οποίο για μας, για το Κοινοβούλιο, είναι καθοριστική σημασία. Δηλαδή, αν θέλουμε να ε, καταστήσουμε τους ελέγχους ε, πιο αυστηρούς, οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν κενά και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά που θα αποφασίσουμε θα εφαρμόζονται κιόλα. Τι να τους κάνουμε τους ελέγχου, όσο καλή και αν είναι, αν σε τελική ανάλυση αυτή που κάνουν τους ελέγχους δεν είναι αποτελεσματική. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Κομισιόν. Αλλά για να το κάνει και αυτό η Κομισιόν πρέπει να έχει μια υποδομή. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου δηλώνονται κάποια προβλήματα, μετά όμως δεν υπάρχει συνέχεια γιατί κανείς θεωρεί ότι δεν είναι αρμόδιος ή γιατί δεν ταιριάζουν τα συστήματα. Ως εκ τούτου ο έλεγχος ε, του ελέγχου και των ελεγκτών θα πρέπει να είναι αποτελεσματικότερος γιατί σε τελική ανάλυση αυτά είναι τα θεμέλια στα οποία μπορεί να βασιστεί να βασιστούν οι οικολογικές καλλιέργειες και επ' αυτού περιμένουμε τις αντιδράσεις της για το πώς μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Με λίγα λόγια, αυτά είχα να σας πω. Έχουμε ακόμα δύο τριμερείς διαλόγους. Ο επόμενος προβλέπεται για την 3η Μαΐου και στις 31 επίσης θα είναι ο άλλος. Είχαμε τις συνεδρίες των συντονιστών, καθορίσαμε εκεί τις ε, προτεραιότητές μας έτσι ώστε στον ε, τελικό τριμερή διάλογο ε, να έχουμε και τον Επίτροπο ενδεχομένω για να καταστεί σαφές το πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά για μας. Είμαι απόλυτα σαφής. Με τη νέα Προεδρία, το να ξαναξεκινήσουμε και όλη αυτή τη διαδικασία να την δρομολογήσουμε από την αρχή, νομίζω ότι αυτό δεν εξυπηρετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και κανέναν άλλο. Ως εκ τούτου πρέπει να το κλείσουμε το θέμα και είμαι αισιόδοξο ότι θα τα καταφέρουμε, διότι νομίζω ότι και η Προεδρία συνειδητοποίησε ότι θα πρέπει να σκεφτεί πίεση και να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το να μην υπάρξει κανένα αποτέλεσμα, αυτό θα ήταν ε, ε, καταστροφή, ε, διότι σας λέω ότι θα πρέπει να, σε εισαγωγικά τώρα, λισαβονοποιήσουμε την νομοθεσία. Πρέπει να επεξεργαστούμε τον κανονισμό για τις οικολογικές καλλιέργειες και σας λέω και πάλι ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Λίντς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την πολύ πλήρη παρουσίασή του σαν σκιώδης Συζητήσαμε για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων μετά από τον τελευταίο τριμερή διάλογο και λάβαμε την πλήρη ενημέρωση. Νομίζω ότι τουλάχιστον μετά τον τελευταίο τριμερή διάλογο με τον συνάδελφο, τον κύριο Χόισλινγκ, Δεν προχωρήσαμε αρκετά και η Προεδρία της Μάλτας νομίζω τουλάχιστον σε αυτή την νέα προσπάθεια και τη συντακτική ομάδα θέλησε να προχωρήσει το θέμα με άλλους ρυθμούς. Υπάρχει αυτή η συμβιβαστική πρόταση. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο θα έλεγα. Και ελπίζω θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πριν το τέλος αυτής της ε, Προεδρίας. Έχουμε κάνει πάντως σημαντικά βήματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και αυτή η νέα πρόοδος, ε, ο νέος κανονισμός να είναι πραγματικά ένα ποιοτικό βήμα για το θέμα αυτό που μας απασχολεί σήμερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σα για μια ακόμη φορά στα βιολογικά θερμοκήπια των σκανδιναβικών χωρών. Και ο φίλο μέλο της Επιτροπή Γεωργίας να επισημαίνω τι ιδιαιτερότητες αυτών των θερμοκηπίων. Ε, θα επιστρέψω στη Λαπωνία και εξακολουθούμε να έχουμε ένα μέτρο χιόνι εκεί. Πάντως η βιολογική γεωργία στη Φιλανδία ε, είναι πολύ πιο παλή από τη νέα κατάσταση και οι πολιτικές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν τροποποιήσει και τον τρόπο ανάπτυξης γεωργικής δραστηριότητας. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Επιτρόπο την Κομισιόν και τον κύριο Χόισλιν που ε, συμφωνούν με τη μνήα της ιδιαιτερότητας των σκανδιναβικών χωρών και των βαλτινικών χωρών και προσφέρουν εξαιρέσεις ε, στις χώρες αυτές που μπορούν να συνεχίσουν τη βιολογική παραγωγή τους σε θερμοκήπια. Βέβαια δεν έχουμε επιτύχει ακόμη το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί προτείνεται υποστρώματα αυτά να περιλαμβάνουν 80% χώμα από τις τοπικές γεωργικές καλλιέργειες, ενώ στα σκανδιναβικά θερμοκήπια χρησιμοποιούν το καλύτερο χώμα που έχουν στη διάθεσή τους, το καλύτερο έδαφος και το πιο κατάλληλο για την καλλιέργεια, χωρίς ε, μάλιστα ε, λιπάσματα. Και τέτοιου είδους ε, υποστρώματα δεν τα χρησιμοποιούμε, δεν τα βρίσκουμε εύκολα αλλού, ούτε καν σε άλλες περιοχές της ίδιας χώρας. Και αν υιοθετηθεί η τελευταία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα φανιστεί η βιολογική παραγωγή σε θερμοκήπια των σκανδιναβικών και βορείων χωρών. Ελπίζω να σημειώσουμε πρόοδο και ελπίζω να λάβετε υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτές της σκανδιναβικής βιολογικής παραγωγής στον τριμερή διάλογο ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε βιολογικά στα θερμοκήπια, στι σκανδιναβικέ χώρε και στι χώρε τη Βαλτική. Δεν νομίζω κανένα εδώ να θέλει να σταματήσει η βιολογική παραγωγή οπουδήποτε στην Ευρώπη. Γιατί κάτι τέτοιο αντιβαίνει στι ίδιε αρχέ τη κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εγώ, ξέρετε, ομιλώ καταρχήν αντικαθιστώντας ε, τον συνάδελφό μου που δεν μπόρεσε να έρθει. Μου έχει γράψει βέβαια αυτά που θέλω να πω. Ο οικολογικός ε, κανονισμός ε, είναι ένα κάτι πολύ περίεργο που αφορά πολλούς ε, τομείς της ε, γεωργίας. Ε, ξέρει ο συνάδελφός μου ότι σήμερα υπήρξε μια μακρά συζήτηση στο επίπεδο των συντονιστών. Τώρα έχουμε φτάσει στην τελευταία φάση στις συζητήσεις με την Μαλτέζικη Προεδρία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την έκθεση και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ε, η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι έτοιμη να καταβάλει επιπρόσθετες προσπάθειες για τις διαπραγματεύσεις και επίσης είναι ακράδαντα πεπισμένη ότι οι τεχνικές συναντήσεις είναι απολύτως απαραίτητες έτσι ώστε στις 3 και στις 31 Μαΐου να προχωρήσουν οι τριμερείς διάλογοι. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να παρακαλέσουμε τη Μαλτέζικη Προεδρία να διαθέτει περισσότερο χρόνο για τις προκατρακτικές συζητήσεις ε, ε, ο πρόεδρος και όλοι οι αρμόδιοι έχουν πει, όπως και ο επίτροπος, ότι μπορούν να συμμετέχουν συναντήσεις ε, ε, μέρους λοιπόν αυτών των αρμοδίων θα ήθελα να πω τρία θέματα. Σπόροι, εκεί επί των σπόρων εξακολουθεί να υπάρχουν συζητήσεις και σε σχέση με το ετερογενές υλικό. Κατόπιν θερμοκήπια, προτινόμενη ζώνη α, αφορά έξι χώρες Βαλτικής, βόρειες χώρες, αυτή η ζώνη μπορεί να λειτουργήσει, όμως το θέμα από πού προέρχεται η γη ε, στις περιοχές αυτές, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Επόμενη λέξη κλειδί, τράπεζα δεδομένων. Και εκεί έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά σε τελική ανάλυση αυτή η πρόοδος είναι συνάρτηση των σπόρων. Όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, πράγματι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να βρούμε λύση επ' αυτού. Ε, Κατόπιν ο συνάδελφός μου αναφέρει ποια βήματα πρέπει να γίνουν και λέει καταλήγοντας ότι θα πρέπει να πείσουμε τη Μαλτέζικη Προεδρία να συμμετέχει σε περισσότερες προκατρακτικές συναντήσεις. Να συμμετέχουν και οι συνεργάτες των πολιτικών ομάδων, αν κρίνεται απαραίτητο, όπως επίσης και οι συγητές. Ε, επίσης, ο συνάδελφός μου ε, παρακαλεί να υπάρξει επέκταση της ομάδας. Δεύτερον, οι συναντήσεις των σχεδόν συγητών θα πρέπει να ε, λάβουν χώρα μετά την 3η Μαΐου για να αξιολογηθεί η πρόοδο και πριν από την 31η Μαΐου έτσι ώστε να μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι δύο συναντήσεις. Και τρίτον ε, πρέπει ε, να προγραμματιστούν ήδη τώρα οι συναντήσεις για να διασφαλίσουμε τη ε, βέλτιστη εύρυθμη λειτουργία. Και ο συνάδελφός μου καταλήγει, η συνέχεια είναι κάτι καθοριστική σημασία και υπογραμμίζει, εμείς επισημαίνουμε, ο εισηγητής να συνεχίσει τη συζήτηση μέχρι τον τελευταίο τριμερή διάλογο όπου όπου ο Επίτροπος θα αναλάβουν την διεύθυνση της συζήτησης, ο Επίτροπος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Ευχαριστώ εγώ τον συνάδελφο, αλλά ευχαριστώ και τον εισηγητή και όλους τους άλλους ε, σκιοδησηγητές. Χαίρομαι που δεν είμαι αρμόδια για αυτή την έκθεση, ε, γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκη έκθεση και χαίρομαι που εγώ μπορούσα να περιστώ μόνο στο να παρουσιάσω την έκθεση αυτή. Ο κύριος Άγνιο. Για μία ακόμη φορά ξαναμιλούμε για τις ε, ευρωπαϊκές διατάξεις για τη βιολογική παραγωγή. Θυμάμαι ότι πριν από τρία χρόνια και παραπάνω ξεκινήσαμε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία κατε, καταγγέλλοντας την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Περιοχής να ρυθμίσει τα πάντα και τα εμπόδια στα οποία προσέκλωσε στο Συμβούλιο. 28 Υπουργοί Γεωργίας στο Συμβούλιο αναγνώρισαν ότι αυτός δεν είναι τομέας ε, κατάλληλος για ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και μάλιστα ο κ. Στάκουλα από τη Φιλανδία, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε ότι οι Φιλανδοί βιολογική παραγωγή, ε, καταναλωτές μάλλον, πολύ ευχαρίστως αγοράζουν βιολογικά οποροκυπευτικά από τα θερμοκήπια της Σκανδιναβίας, παρόλο που γίνεται εισαγωγή ε, του χώματος, γιατί δεν τους ενδιαφέρει τους καταναλωτές, είναι πολύ ικανοποιημένοι με τα προϊόντα που αγοράζουν. Οπότε φαντάζομαι ε, δεν θα πούνε οι καταναλωτέ Φιλανδία στον ε, Φιλανδό Γεωργό ότι δεν τηρεί τους κανόνες. Δεν υπάρχει καμία ε, αίτηση από πλευρά καταναλωτών για ρύθμιση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, αν ρωτήσουμε έναν ε, τυπικό αγοραστή καταναλωτή, βιολογικών προϊόντων, που είναι 4% πανευρωπαϊκά, και του ρωτήσουμε τι περιμένει. Καταρχήν είναι κατά των, της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων στις βιολογικές καλλιέργειες, δεν θέλουν λιπάσματα. Επίσης δεν θέλουν συνθετικά ή ε, χημικά παρασιτοκτόνα και φυτοφάρμακα και επίσης θέλουν ε, στη βιολογική κτηνοτροφία να είναι ελευθέρας βοσκής ε, τα ζώα. Αυτά είναι τα βασικά τρία χαρακτηριστικά που περιμένουν οι αγοραστές βιολογικών προϊόντων. Τώρα, αν θέλετε να ρυθμίσετε την παραμικρή λεπτομέρεια και να έχετε μια ενορμανισμένη διαδικασία σε 28 χώρες μέλη, θα κάνετε το βίο αβίωτο στους ε, βιολογικούς παραγωγούς. Οπότε θα τους οδηγήσετε σε αβαριφαρισμό ή θα ε, εξακοντήσετε σε αστρονομικές τιμές τα βιολογικά προϊόντα με τις τόσο υπερβολικές απαιτήσει. Να αφήσετε λοιπόν τις ρυθμίσεις αυτές στου πιστοποιημένου στους πιστοποιημένους στα επιμέρους κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να επανέλθω στα θέματα των καταλήπων των φυτοφαρμάκων. Σε σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται και κανένας καταναλωτής δεν καταλαβαίνει εδώ να γίνουν αυστηρότερα ακόμα τα όρια. Παραδείγματος χάρη στο Βέλγιο βλέπουμε ότι αυτό το 0,1 μικρογραμμάριο ανά κιλό, που είναι το όριο που έχει θετηθεί και ακούω μάλιστα και αυτή είναι και η ερώτηση που θέλω να κάνω στον εισηγητή αν θα μπορούσε να υπάρξει ένα συμβιβασμός, δηλαδή να αφαιθεί αυτό το θέμα για τα κράτη-μέλη να το αποφασίσουν. Πιστεύω ότι εδώ αν υιοθετήσουμε αυτήν, την, αυτό το όριο θα είναι η χειρότερη λύση. Και παραδείγματος χάρη σε μένα στη δική μου περιοχή τα οποροκυπευτικά για τα μήλα παραδείγματος χάρη τα οποία ενδεχομένω θα εισάγονται χωρίς απολύτως κανένα ε, τέτοιο φυτοφάρμακο κατάλοιπο δεν θα μπορούν σε σχέση με την εσωτερική παραγωγή να ανταποκριθούν σε καμία περίπτωση. Νομίζω λοιπόν ότι αν κοιτάξει κανείς σήμερα τους αριθμούς που έχουμε και μετά από εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους και αναλύσεις βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση. Ξεπερνούν, τουλάχιστον στη δική μου περιοχή, και σας μίλησα για τα οποροκυπευτικά, για τα μήλα και για τις βιολογικές ε, καλλιέργειες, ξεπερνούν αυτά τα όρια και δεν έχουμε καμία απολύτως ε, ε, από τους ελέγχους που κάναμε αποδείξεις ότι ξεπερνούνται αυτά τα όρια. Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που ένα, σε έναν έλεγχο, ένα και μοναδικό μήλο ξεπεράσει αυτά τα όρια, σε αυτή την περίπτωση όλη η παραγωγή όλης της περιοχής αυτής δεν θα μπορεί να πιστοποιείται σαν βιολογική και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί η συμβαστική λύση εδώ. Δύο πράγματα λοιπόν θα γίνουν. Είτε θα αλλάξει αυτό το όριο, είτε θα πρέπει κάθε φορά που ελέγχεται μία παραγωγή να αφήνεται το όριο. Δεν θέλω, κατά την άποψή μου, δεν θέλω να υιοθετηθεί αυτό το, αυτός ο κανονισμός, γιατί κανείς δεν θα μπορεί μετά να εξηγήσει πώς θα είναι δυνατόν ένα βιολογικό προϊόν να μπορεί να έχει τα ίδια κατάλοιπα, τα ίδια όρια, όπως και ένα συμβατικό φρούτο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δείξουμε καλή θέληση, λογική, την κοινή λογική και για μένα το καλύτερο, το καλύτερη συμβαστική λύση εδώ θα ήταν να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τις μεθόδους και του ελέγχου και να μην επιβάλλουμε τόσο αυστηρές τιμές που να μην μπορεί κανείς να τις στηρίσει. Ευχαριστώ κύριε Στάκολα. Ευχαριστώ. Μια και έχουμε διερμηνή από τα φιλανδικά, θα ήθελα κι εγώ να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Γιατί ε, μου λένε πολύ ότι είναι πολύ δύσκολα τα φιλανδικά και θέλουν, χρόνια ολόκληρα για να τα μάθει κανείς. Ε, εν πάση περιπτώσει, ο κύριο Άγνιου αναφέρθηκε προσωπικά σε μένα και μου λένε ότι όταν γίνονται προσωπικά σχόλια οφείλουμε να απαντήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν πώ θα εφαρμόσουν την οδηγία. Θα πρέπει να είναι αρκετά ελαστική οδηγία και να του επιτρέπει τέτοια διακριτική ευχέρεια. Επίση, ε, όταν μιλούμε για βιολογική γεωργική παραγωγή και κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη που δεν υπάρχει ε, βιομηχανία δεν υπάρχει χημική βιομηχανία. Το έδαφος είναι ελεύθερο από τη μόλις από χημικά προϊόντα και μιλούμε μάλιστα και για ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές ε, με τη φύση να είναι πεντακάθαρη και απαραγμένη από τη ρήπαση. Πιστεύω ότι και ο φυλαδός καταναλωτής αλλά και ο Ευρωπαίος καταναλωτής γνωρίζει ότι η φυλαδική αυτή η βιολογική παραγωγή είναι απόλυτα καθαρή. Βέβαια, δεν έχουμε καταφέρει να πουλήσουμε τα προϊόντα μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά είναι ενδιαφέρον που τελικά νομίζω όλοι οι συνάδελφοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να προβλέψουμε αρκετό περιθώριο λιγμών ε, και ελαστικότητα στην εφαρμογή της οδηγίας για να μπορέσουμε να θέσουμε σε εμπορία και τα φιλανδικά βιολογικά προϊόντα που είναι συνώνυμα υγιεινών, καθαρών ε, και αγνών προϊόντων. και μάλιστα έχουμε πολύ αποδοτική παραγωγή απορροκυπευτικών. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα επανέλθω λιγάκι σε αυτό το θέμα, διότι ξέρετε κάτι, είπαμε αρκετά αυστηρά ότι κατ' ουσίαν αυτά, θα πρέπει να ισχύουν για τις ε, ε, εκμεταλλεύσεις που είναι των 20 εκταρίων και που το ήδη πράττουν. Όταν όμως έγινε συζήτηση ξαφνικά τι είπαν, είπανε ότι ε, όλοι θα μπορούν να το πράττουν αυτό όσοι θέλουν να έχουν ανεξάρτητη παραγωγή. Άρα δηλαδή τίθεται το ερώτημα θα προστατεύσουμε τους παραγωγούς εκείνους που έτσι και αλλιώ έχουν προβλήματα ε, λόγω των καιρικών συνθηκών ή ε, θα επιτρέψουμε όλα αυτά τους ανεξάρτητους γεωργούς ανεξαιρέτως και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει κάποιες, ε, κάποιες τρευλώσεις ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ιταλία και άλλες χώρες. Πρέπει να είμαστε πιο περιοριστικοί. Ζητήσαμε τον, τον ε, συμβασμό ε, προσπαθήσαμε να ορίσουμε τις ε, περιφέρειες πρέπει πράγματι να ξεκαθαρίσουμε από πού θα προέρχεται το χώμα. Πρέπει όμως και να περιορίσουμε τις εξαιρέσεις, γιατί αλλιώς ξέρετε κάτι, θα έχετε ανταγωνισμό από άλλους παραγωγούς ε, και ε, αυτό θα ήταν μια εκτενέστατη ερμηνεία. Μέσα στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, ε, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι υπάρχουν ειδικέ μέθοδοι παραγωγής, εμείς θα θέλαμε να είμαστε πιο περιστικοί, να υπάρχει δυνατότητα περισσότερων εξαιρέσεων, αλλά δυστυχώς ε, λόγω της πλειοψηφία ε, στο Συμβούλιο δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Αγαπητέ συνάδελφο Ντόρφμαν, σχετικά με τα φυτοφάρμακα, πρόκειται ακριβώς από αυτού. Και εγώ τη γνωρίζω αυτή τη μελέτη και εμείς ε, την κάναμε στη Γερμανία σχετικά με το από πού προέρχονται τα φυτοφάρμακα, ε, μπορεί κανείς να πει ότι κατ' ουσίαν αυτό είναι ένα θέμα που αφορά ε, τον γείτονα, γιατί υπάρχουν ε, περιοχές καλλιέργειας τροφίμων και φρούτων, όπου τα φυτοφάρμακα δεν παραμένουν σε ένα μόνο σημείο, μεταφέρονται. Ως εκ τούτου ε, δεν μπορούμε να πούμε τώρα στους ε, ε, βιοκαλλιεργητές ότι ξέρετε εσείς δεν μπορείτε να πουλάτε τα προϊόντα σας γιατί αν το κάνουμε αυτό ε, θα τους καταστρέψουμε. Και πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της Κομισιόν η οποία Παραδείγματο χάρη σε άλλε περιπτώσει, όταν επρόκειτο για τι βρεφικέ τροφέ, ε, σκόντεψε να καταστρέψει σχεδόν μία ολόκληρη επιχείρηση. Το λέω λοιπόν για άλλη μια φορά, ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, κανονισμοί είτε για την απόσταση είτε για τι εξασφαλίσει και ε, μετά μπορούμε να τα συζητήσουμε με την ησυχία μας. Βεβαίως η δική μας η πρόταση είναι τώρα και γι' αυτό δεν είμαι ευτυχής με την πρόταση του Συμβουλίου ε, που λέει το Συμβούλιο ότι κάθε χώρα να κάνει ό,τι θέλει, να μην έχει κανονισμούς. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να πούμε ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που επιθυμεί και ξέρετε τι επιθυμούμε. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν εναρμονισμένες προδιαγραφές στην Ευρώπη ε, χωρίς στρέβλωση ανταγωνισμού. Ε, αν όμως αυτές οι τρεις χώρες συνεχίσουν να καταψηφίσουν το Συμβούλιο θα αναγκαστούμε και εμείς να βρούμε κάποια άλλη λύση. Η δική μας πρόταση είναι να μην προσθεθούν και άλλες χώρες αλλά αυτές που επιτρέπεται να το πράττουν, οι τρεις αυτές ε, να παραμείνουν οι μόνες και μετά οι υπόλοιποι να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή ε, το Συμβούλιο είναι διαιρεμένο. Εάν δεν περάσει αυτή η πρόταση στο Συμβούλιο θα απορριφθεί το σύνολο του πακέτου ε, της δέσμης μέτρων. Και ξέρετε ότι και στο Κοινοβούλιο μέσα στις πολιτικές ομάδες υπάρχει διάσταση απόψεων, άρα δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πρώτα τα δεδομένα και μετά νομίζω ότι θα μπορέσουμε πολύ συγκεκριμένα και αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Σας το λέω όμως και πάλι με απόλυτη σαφήνεια, αν ε, θεωρείτε ότι ε, δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή κυρίως των κονδυλίων που προβλέπονται για τις οικολογικές καλλιέργειες, τότε θα πρέπει να αντιδράσουν τα κράτη-μέλη δεν θα επιτρέπεται, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρονται τα φυτοφάρμακα χιλιόμετρα ολόκληρα. Το έχω πει επανειλημμένα και στις πρώτες συζητήσει. Η μόλυνση, η ρήπανση μάλλον από τα φυτοφάρμακα δεν οφείλεται στις οικολογικές καλλιέργειες. Δεν μπορεί κανείς να φορτώσει τα πάντα σε οικολογικέ καλλιέργειε. Γιατί αν έτσι τελικά οικολογικέ καλλιέργειε θα έχουμε μόνο στη Λαπωνία. Στο Τυρόλο α πούμε αποκλείεται να υπάρχει οικολογική καλλιέργεια. Όμω, σε τελική ανάλυση, εφόσον υπάρχει το δικαίωμα συμβίωση για όλου του πολίτε υπάρχει και για τους καλλιεργητέ. Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Αν θέλετε και οποτεδήποτε θέλετε, μπορείτε να έρθετε να με βρείτε Έχουμε ακόμα συναντήσεις και οδών εισηγητών, έτσι ώστε οι συμβασμοί που θα υποβάλουμε να έχουν συζητηθεί εκ των προτέρων με τους εισηγητές. Δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά τι να κάνουμε, πολλές φορές κάποιοι θα πρέπει να δέχουν την άποψη της πλειοψηφία. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Ολοκληρώσαμε η συζήτηση. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση, ακούσαμε και τις απαντήσεις του εισηγητού. Ελπίζω να καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε το θέμα αυτό με τους τριμερείς διαλόγους ε, κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας. Περνάμε στο επόμενο σημείο, στις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Eurostat που θα μας παρουσιάσει την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, και το έγγραφο 0786 του 2016 μετά την επισκόπηση για τη δομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που υπάρχει από το 1966 και εξασφαλίζει εναρμονισμένα στοιχεία και δεδομένα για τη δομή των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και μια απογραφή που γίνεται περίπου κάθε 10 χρόνια και μάλιστα περιλαμβάνει πολλά στοιχεία όχι μόνο για το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το είδος της γεωργικής δραστηριότητας, αλλά αφορούν και άλλα πολύ πολυάριθμα στοιχεία, όπως είναι κάποιες μη γεωργικές οικονομικές δραστηριότητες που γίνονται επί της γεωργικής εκμετάλλευσης. Το σύστημα μάλιστα αυτό της επισκόπησης δομή γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί την ραχοκοκαλιά του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, Γεωργικών Στατιστικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα ένα νέο σύστημα πιο ελαστικό ε, που θα αντικαταστήσει τον κανονισμό 1166 του 2008. Η κυρία Κριστίν Βίρτς θα μας κάνει την εισαγωγή εκ μέρους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το οποίο είναι η συγκέντρια κυρία Νταντσίλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Κριστίνα Βίρτς, είμαι αναπληρώτρια Γενική Διευθυντρία για Περιφερειακές ε, και ε, τοπικές ε, στατιστικές ε, και γεωργικές στρατηγικές στην Eurostat. Και χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πλαίσιο κανονισμού για τις ενοποιημένες στατιστικές γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Όπως είπατε και εσείς, εδώ και 60 χρόνια τώρα η Eurostat και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τις, ευρωπαϊκές, με τις στατιστικές υπηρεσίες παρέχουν μια σειρά στοιχείων γεωργικών ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την πολιτική που στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά και μάλιστα ε, περιλαμβάνουν στοιχεία για τη ε, γεωργική στρατηγική, για τις περιβαλλοντικές δράσεις που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αξιόπιστες και συγκρίσιμες ε, γεωργικές στατιστικές πληροφορίες που θα πρέπει όμως να προσαρμόζονται και σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο για να είναι εύχριστα γιατί και η παγκόσμια γεωργία και το παγκόσμιο κλίμα αλλάζει, αλλά και οι επίσημες στατιστικές αλλάζουν. Αυτή τη στιγμή ε, οι ευρωπαϊκές γεωργικές στατιστικές στηρίζονται σε ένα κατακαιρματισμένο σύστημα με νέα ε, βασικές δράσεις ε, και μεγάλο άχθος για τη συγκέντρωση των στατιστικών, ενώ οι ανάγκες στοιχείων αυξάνονται και για την κοινή γεωργική πολιτική και για άλλες πολιτικές, ενώ οι πόροι μας συρρυκνώνονται. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε τη νομική βάση για διαρθρωτικές στατιστικές πληροφορίες και κάθε δεκαετία ε, πραγματοποιούμε και απογραφές γεωργικές και μάλιστα η νομική αυτή βάση εξέπνευσε το 2016 ε, για τη βάση δεδομένων, οπότε έχουμε γεωργική ε, Απογραφεί όχι μόνο κάθε 10 χρόνια, αλλά και διάμεσες ε, απογραφές, δειγματοληπτικές ε, ε, κυρίως κάθε τρία-τέσσερα χρόνια. Είναι κατακαιρματισμένο λοιπόν αυτό το νομικό πλαίσιο και τώρα πια δεν έχουμε καν νομική βάση για την επόμενη γεωργική απογραφή. Γι' αυτό και έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική γεωργικών στρατηγικών ε, από το 2020 και παραπέρα. Πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο σύστημα για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών γεωργικών στατιστικών θέλουμε να, να ικανοποιήσουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές μας στατιστικές ανάγκες και να κρατήσουμε το άκθος και το κόστος υποέλεγχο για τα Εθνικά Ινστιτούτα Στατιστικής αλλά και για τους Ευρωπαίους Γεωργούς. Ε, αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι μια ε, διπλή προσέγγιση σε δύο φάσεις με δύο ε, κανονισμούς πλαίσιο. Ο πρώτος εξασφαλίζει το, τη γεωργική απογραφή και τα διαφορετικά δεδομένα σε επίπεδο μεμονωμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συγκεντρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία στο δεύτερο κανονισμό πλαίσιο. Τα τελευταία δύο χρόνια, από το 2013 συγκεκριμένα, έχουμε αναπτύξει τον πρώτο κανονισμό πλαίσιο για τις ενοποιημένες στατιστικές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτόν θα σας παρουσιάσω σήμερα. Θα ήθελα μάλιστα συντομία να σας παρουσιάσω πώς ο κανονισμός αυτός ε, για τις ενοποιημένες στατιστικές γεωργικών εκμεταλλεύσεων, IFS, ε, συγκεντρώνει διαρθρωτικές πληροφορίες σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και επιτρέπει την συμπερίληψη ε, της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής διάστασης της γεωργίας τα στοιχεία αυτά. Για παράδειγμα, ε, μας επιτρέπει την αξιολόγηση του αντικτύπου κάποιων πολιτικών και την ανάλυση τους ανα ε, ε, γεωργικής εκμετάλλευσης, ε, ηλικίας, ε, μεγέθους ε, γεωργικής εκμετάλλευσης ή συνδυασμό των άνω χαρακτηριστικών. Όπως είπα, θα ακολουθήσει δεύτερος κανονισμός πλαίσιο αργότερα και θα καλύπτει αιτήσει στατιστικές για κτηνοτροφική και γεωργική παραγωγή, ε, προμήθεια σπόρων, ε, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη γεωργία, καθώς και τα πρώτα βήματα της μεταποίησης, μετά τη γεωργική εκμετάλλευση δηλαδή, και κυρίως για τα ζωικά προϊόντα, όπως είναι σε σφαγεία, σε γαλακτοκομικές μονάδες και επίσης ε, ε, θα έχουμε και κάποια στατιστικά στοιχεία για τη βιολογική παραγωγή. Για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τόσο σημαντική πολιτική όπως είναι αυτή για τη βιολογική παραγωγή που συζητήσατε πριν από λίγο. Τώρα, ποια είναι η δομή του νέου κανονισμού για τις ενοποιημένες στατιστικές. Καταρχήν έχουμε μία ομάδα κρίσιμων δεδομένων που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες τις εκμεταλλεύσεις που έχουν ένα ελάχιστο μέγεθος, ελάχιστες διαστάσεις. Και αυτό έχει μία πτυχή την έκταση, τη, το ζωικό κεφάλαιο και τη διαχείριση, δηλαδή το, τον ποιο λαμβάνει αποφάσει για τη λειτουργία τη γεωργική εκμετάλλευση. Και τέτοιε πληροφορίε θα τι λαμβάνουμε από όλε τι γεωργικέ εκμεταλλεύσει που περιλαμβάνονται στην απογραφή και τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται σε αυτή τη βασική πράξη που θα σα υποβάλουμε, αυτόν τον κανονισμό πλαίσιο. Και αυτές οι πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε θα συμπληρώνονται και από κάποια άλλα τμήματα, από δομές που θα έχουμε στο πρόθεσμό χρονικό ορίζοντα, γιατί δεν θα χρειαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές ε, ε, ετησίως. Για παράδειγμα, για τις δομές των οπορώνων ε, ή των αμπελιών Επίση έχουμε κάποια στοιχεία για τις ε, πρακτικές διαχείρισης του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στη γεωργική εκμετάλλευση, αλλά και κάποια περιβαλλοντικά στοιχεία όπως θα είναι η διαχείριση των, λοιπασμάτων, του εδάφους, ε, ε, αγροτική ανάπτυξη, άρδευση και ούτω καθεξής. Και όλα αυτές, όλες αυτές οι πληροφορίες θα συγκεντρώνονται μόνο από ένα μικρό δείγμα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όχι όλων αυτής της απογραφής και όχι ταυτόχρονα. Έτσι, το, το άχθος του, του κανονισμού οι διατυπώσεις θα είναι λιγότερο βαριές από ό,τι στο παρελθόν. Το νομικό πλαίσιο προβλέπει αυτά τα επιμέρους τμήματα και επιμέρους κατηγορίες να καθορίζονται στον κανονισμό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά να προσδιορίζονται σε εφαρμοστικούς κανονισμούς. Έτσι θα έχουμε την απαραίτητη ελαστικότητα ώστε να προσαρμόσουμε ε, και χρονικά την συγκέντρωση των δεδομένων, αλλά και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε κατάλληλα τις πολιτικές μας και να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες ε, διοικητικές πηγές δεδομένων για να συμπληρώσουμε τις ανάγκες μας σε δεδομένα. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης την εισαγωγή ad hoc απογραφών ε, για συγκέντρωση δεδομένων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει και αυτή τη δυνατότητα ώστε αν ανακύψουν νέα στοιχεία, νέα ζητήματα σε πολιτικές, στη νέα κοινή γεωργική πολιτική, που θα γίνουν γνωστά αφού προσδιοριστεί και η νομική βάση για την συλλογή των δεδομένων, τότε θα προσδιοριστούν και νέες συλλογές δεδομένων και αυτό μέσω των εφαρμοστικών κανονισμών. Η προτινόμενη χρήση εφαρμοστικών και καταξιοδότηση πράξεων εξασφαλίζουν την ε, απαραίτητη ελαστικότητα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα, στη ζήτηση δεδομένων ε, από τους ηθήνοντες των πολιτικών. Θεωρούμε ότι αυτή η ευελιξία είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται, η ψηφιοποίηση εντείνεται και αν πρέπει τώρα να καταγράψουμε τι ε, μεθόδους παραγωγής δεδομένων θέλουμε να καταγράψουμε για το μέλλον. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι ώστε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στις μελλοντικέ ανάγκες. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος κανονισμός πλαίσιο για τις ενοποιημένες στατιστικές και προβλέπει ότι η γεωργική απογραφή μπορεί να γίνει το 2020 και να ακολουθήσουν δειγματοληπτικές έρευνες το 2023 και το 2026. Αυτός ο κανονισμός μάλιστα πλαίσιο θα απαλλάξει τους γεωργούς από τις υπερβολικές ε, διατυπώσεις και σε μερικές χώρες μέλη θα μειώσει και τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που καλύπτονται από την απογραφή θα μειωθούν στο μισό, για παράδειγμα, οι γεωργικές εκμεταλλευσει που θα εμπλακούν στην απογραφή στη Μάλτα και τη Ρουμανία. Και μάλιστα μέχρι το 2020 3,5 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν θα εμπίπτουν στην απογραφή με βάση τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να υλοποιήσουμε λοιπόν αυτό το στόχο και να πραγματοποιήσουμε γεωργική απογραφή στην Ευρώπη ώστε να καταλήξουμε σε συγκρίσιμα δεδομένα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το 2018, ώστε να έχουν το χρόνο τα κράτη-μέλη να ετοιμαστούν μέχρι το 2020, γιατί ε, χρειάζεται αρκετή δουλειά και προεργασία. Σε σύγκριση με το παρελθόν πάντως, ο νέος κανονισμός προβλέπει νωρίτερη παροχή των δεδομένων σε σχέση με προηγούμενες απογραφές, ώστε να χρησιμοποιούνται εγκαίρως για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες πολιτικής. Αυτά και είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε το νέο κανονισμό πλαίσιο για τις ενοποιημένες στατιστικές της γεωργικής εκμεταλλεύσης με τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Σας ευχαριστώ κύριο Στάκουλα. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για τις προτάσεις που μας παρουσίασε να πω κι εγώ δύο λόγια εκ μέρους της ομάδας των ε, φιλελευθέρων. Η συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη γεωργία είναι πολύ σημαντική, διότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση και μπορούμε να εντοπίσουμε δυσκολίες, προβλήματα και να έχουμε και μια καθοδήγηση όσον αφορά τις προτινόμενες αλλαγές και τις πολιτικές που αφορούν ε, τους γεωργούς και τη γεωργία. Είναι σημαντική για τις ε, αγρότες τους ίδιους, αλλά και για την ανάλυση από μέρους των ε, οργανώσεων των παραγωγών για την κατάσταση στη γεωργία για την καινοτομία και τις νέες ε, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Θα συζητήσουμε αλλαγές στους ε, κανόνες που διέπουν τις εναρμονισμένες στατιστικές. Η βάση είναι το 1996. Οι νέοι κανόνες θα χρησιμοποιηθούν για την ε, νέα γεωργική απογραφή που θα λάβει χώρα το 2020. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε τους κανόνες αυτούς το συντομότερο δυνατόν για να είμαστε έτοιμοι για αυτή την ε, γεωργική απογραφή του 2020. Την ίδια ώρα θα πρέπει να έχουμε τις καθευθυντήριες γραμμές να αποφύγουμε επιπλέον ε, ε, δουλειά και άχθος για τους ίδιους τους γεωργούς όσον αφορά τη συλλογή αυτών των στοιχείων τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τις αλλαγές ε, στην κατάσταση των γεωργών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι στατιστικές θα με τον πιο οικονομικό τρόπο και ότι θα ενσωματωθούν ε, στον σχεδιασμό και στην καθημερινή τους ε, δουλειά. Αυτό το βλέπουμε εξάλλου και στις προτάσεις της ομάδας που δημιουργήθηκε για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε αυτοί οι νέοι κανόνες να προετοιμαστούν εγκαίρως για την νέα γεωργική απογραφή, να δημιουργήσουν τα λιγότερα προβλήματα για τους ίδιους τους αγρότες και να καλύπτουν τους περισσότερους δυνατούς τομείς. Πρόεδρε, εγώ θα διαβάσω κάτι. Θα διαβάσω αυτά που μου είπε ο συνάδελφο Βανκασέλ, ε, είναι ο συγητή τη πολιτική μα ομάδα και δυστυχώ δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Λέει λοιπόν ότι η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια νέα προσέγγιση ενοποιημένων στατιστικών, στατιστικών συστημάτων για τι γεωργικέ εκμεταλλεύσει έχει ως στόχο να έχουμε ένα συνεπέ και αποτελεσματικό σύστημα στατιστικών δεδομένων. Πρέπει να βελτιωθούν τα δεδομένα και υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εδώ λοιπόν ο κύριος Βαν Κασέλ πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει απλούστευση, καλύτερη ποιότητα των δεδομένων, να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση και παράλληλα να μειωθεί η ε, γραφειοκρατία. Υπάρχουν αυτά στην πρόταση και είναι θετικά. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες, η διαχείριση των δεδομένων, αυτά θα έχουν ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις ε, όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στη γύρω Eurostat και στα νέα κράτη-μέλη. Αυτά είχα να σας πω και σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω μέρους των ε, εισηγητών, των σχεδόν εισηγητών. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει με μεγάλη σοβαρότητα να γίνεται αυτή η συλλογή των στατιστικών στοιχείων που αφορούν την γεωργία και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια, κάτι που ζητούν όλο και περισσότερο και περιμένουν ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πρόκειται για ποσά τα οποία είναι ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσα και τους ε, ε, άλλους εισηγητές. Θα πρέπει όμως να συνεννοηθούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στατιστικά στοιχεία αν ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται ε, είναι ακριβώς αυτός για τον οποίο τελικά θα χρησιμοποιηθούν. Τα τελευταία 50 χρόνια Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες ε, ανισότητες, ε, θα έλεγα και ανισορροπίες στο σύστημα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Είναι λογικά αυτά λοιπόν που διαβάζω εδώ στα παραρτήματα της πρότασης αυτής, αλλά πιστεύω ότι με τους εισηγητές, με τους κοιόδες ε, εισηγητές μαζί, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, παραδείγματος χάρη, θέματα που αφορούν τους νέους γεωργούς, την ηλικία που κάποιο τελικά ξεκινάει αυτή την οικονομική δραστηριότητα, επίσης θέματα που αφορούν τον τύπο του εδάφους, κάτι που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την ανάλυση αυτών που αφορούν το θέματα του δεύτερου πυλώνα. Θέματα επίσης ιδιοκτησιακά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη νέα γενιά των γεωργών, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συλλέξουμε και κάποια προβλήματα που αφορούν την γύραση του πληθυσμού στη γεωργία, θέματα φύλου που αφορούν επίσης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τώρα, το θέμα των ε, προθεσμιών όσον αφορά την υποβολή των στοιχείων, κάτι που αφορά ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πιστεύω ότι η προετοιμασία αυτών των εκθέσεων ε, για το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά σίγουρα εδώ βάσει των νέων απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει σίγουρα να δοθούν κάποιες οδηγίες για τα χρονοδιαγράμματα, τις προθεσμίες, για την υποβολή αυτών των νέων στοιχείων, για την έγκαιρη προετοιμασία των εκθέσεων. Κάτι που επίσης μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία, κυρίως όσον αφορά το κεντρικό θέμα που αφορά σήμερα την ε, γεωργία, δηλαδή τη θέση των αγροτών, τη θέση των γεωργών στην τροφική αλυσίδα. Θα θέλαμε λοιπόν λίγο να τροποποιήσουμε αυτήν την ε, πρόταση. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε επιπλέον ε, γραφειοκρατικό άκθος. Αυτό το επαναλαμβάνω. Έχουμε ήδη κάποιες απαιτήσει όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Εμείς θέλουμε να εμπλουτίσουμε την πρόταση χωρίς να δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, οπότε να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Βίρτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στα σχόλια των Ευρωβουλευτών. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Αλλά δεν είστε και υποχρεωμένοι. Thank you for this first... Σας ευχαριστώ πολύ ε, για τις αντιδράσεις σας ε, στις ε, προτάσεις μας. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση που κατά την άποψή μου μπορεί να εφαρμοστεί αρκετά λογικά από τους γεωργούς και λάβαμε υπόψη μας όλες τις πληροφορίες που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Κατανοώ βέβαια ότι ενδιαφέρεστε να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ε, και με πολύ μεγάλη μας χαρά να συζητήσουμε μαζί σας. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς ε, αποτελεσματική μπορεί να είναι πράγματι η συγκέντρωση δεδομένων. Και θα πρέπει να αποφύγουμε ε, να μην απαντούν οι γεωργοί ε, στην περίπτωση που το ερωτηματολόγιο είναι μακροσκελές. Να θελήσουν να αποφύγουν τις απαντήσεις. Τέλος, όσον αφορά αυτά που ελέγχθησαν για το ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να μεταφέρει και να δίνει περαιτέρω τα δεδομένα. Ξέρετε, εμείς το κάνουμε αυτό το συντομότερο δυνατόν, μόλις έχουμε στη διάθεσή μας ε, καλά ε, ε, δεδομένα από τα κράτη-μέλη. Αλλά όπως σας είπα, με πολύ μεγάλη μας χαρά να τα συζητήσουμε αυτά κατά τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση στις 22-23 Μαΐου όταν θα μας παρουσιάσει η συγγήτρια την έκθεσή της. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο ευχαριστώντας ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και τους συναδέλφους για τη συζήτηση και περνούμε ε, στην έγκριση των ε, συστάσεων της Επιτροπής Άγκρη. Θα σας στείλουμε τις συστάσεις των συντονιστών από την πρωινή συνεδρίαση και με έγγραφο και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Και αν δεν υποβληθούν ενστάσεις θα θεωρηθούν συγκεκριμένα τα πρακτικά. Για τα διάφορα δεν βλέπω τίποτα. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει 2 και 3 Μαΐου. Ολοκληρώσαμε την απογευματινή μας συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και σας εύχομαι καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει και εύχομαι σε όλους καλές γιορτές. Είστε επανειδή. Καλή επιστροφή. Γεια σας.